Κυρία Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται. Έλαβα εκ μέρου των ομάδων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών αιτήσει τροποποίησης στις κοινοβουλευτικές επιτροπές και στις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες ο κατάλογος των διορισμών θα δημοσιευθεί στα συνοπτικά πρακτικά αυτής της Συνόδου. Εάν δεν υπάρξουν παρατηρήσεις ως προς την, ε, ως προς την έγκριση των συνοπτικών πρακτικών, οι διορισμοί θα εγκριθούν. Συνεχίζουμε την ημερήσια μας διάταξη, η οποία προβλέπει απόψε την προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την κύρωση και την εφαρμογή των αναθεωρημένων συμβάσεων τους διεθνούς οργάνους εργασίας. Ε, θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τους συντάκτες. Το λόγο λοιπόν έχει για τρία λεπτά ο προ... ένας από τους συντάκτες, ο κύριος Σέρκας. Mr. Σέρκας. Gracias, señora presidenta. Buenas noches, colegas. Buenas noches a los miembros de la comisión que nos acompañan. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γνωρίζουμε ότι η παγκοσμιοποίηση, η οικονομική κρίση και οι μελλοντικέ προκλήσεις σημαίνουν ότι πρέπει να προσεγγίσουμε τα πράγματα παγκοσμίω. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται μόνο μια εθνική και περιφερειακή προσέγγιση. Γι' αυτό η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΔΟΕ είναι ένα σημαντικό ζήτημα με την τριμερή της μέθοδο, η Διεθνής Οργάνωση Εργασία ε, εκπονεί μια εργασία η οποία σκοπό έχει να ε, εξορθολογήσει τις ε, συνθήκες εργασίας. Εμείς εργαζόμαστε με ένα κοινωνικό μοντέλο και είναι απαραίτητο αυτό αλλιώς θα ήταν σαν να ζούσαμε σε έναν άδικο κόσμο. Θέλουμε απλώς τώρα να πρωταγωνιστήσουμε στη δημόσια σκηνή σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ένωση και τα κράτη-μέλη εργάζονται υπέρ αυτού και υπέρ ε, της ε, πρωτοβουλίας ε, του Διεθνούς Γραφείου Απασχόλησης για να βελτιωθεί η κατάσταση σε ό,τι αφορά την ανεργία. Όμως δεν υπάρχει απαραίτητη συνοχή και συνέπεια μεταξύ αυτό που λέμε εμείς και αυτό που κάνουμε εμείς. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε σήμερα για το θέμα και αύριο να βγει ένα ψήφισμα για την επικύρωση των βασικών νομοθετικών οργάνων της, ε, του Διεθνούς Γραφείου Απασχόλησης. Στην ανακοίνωσή σας για τη νέα κοινωνική ατζέντα απευθύνατε εκ νέου έκκληση στα κρατη τα οποία όμως δεν ανταποκρίθηκαν καλέσατε τα κρατημέλη να επικυρώσουν τις σχετικές διεθνεί ε, συμβάσει. Τώρα πρέπει να κάνουμε κάτι πολύ πιο φιλόδοξο. Τα κράτη-μέλη ε, δεν έχουν επικυρώσει όλες τις συμβάσεις ε, της της, ε, του, Διεθνού Γραφείου, του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, ε, της ε, Διεθνής Οργάνωσης, της Οργάνωσης Εργασίας. Χάνουμε έτσι πολλές ευκαιρίες. Χάνουμε έτσι την δυνατότητα να μεταφράσουμε στην πράξη αυτό που εξαγγέλουμε με λόγια. Δεν είναι το να αρκούμεθα σε ρητορικές μόνο παρεμβάσεις. Γι' αυτό ε, θέλουμε κάτι πρακτικό να προκύψει. Όχι μία έκκληση, μία ανακοίνωση, κάτι πιο, δεν τολμώ να πω αλλά τέλος πάντων κάτι πιο ισχυρό. Είναι θέμα συνέπειας, είναι θέμα αξιοπιστίας. Γι' αυτό ε, το ζητούμε, για να μας πιστέψουν οι πολίτες, για να μας εμπιστευθούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σέρκας. Ο κύριος Χάρκιν έχει το λόγο τώρα για τρία λεπτά έκκλησης συντάκτης. Α, η κυρία Χάρκιν, I'm sorry, I'm sorry, Ms. Χάρκιν. You have the floor. Madam President Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, χαίρομαι που συζητούμε την κύρωση και την εφαρμογή των αναθεωρημένων συμβάσεων της ΔΟΕ από τα κράτη-μέλη όταν δημιουργήθηκε το 1990 η ΔΟΕ ε, αυτό έγινε γιατί πιστεύαμε ότι μία μόνιμη ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν υπάρχουν συν, σωστές συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους. Αγωνίζεται λοιπόν η οργάνωση αυτή για σωστές συνθήκες εργασίας και αξιοπρέπεια σε όλο τον κόσμο. Είναι πολύ καλό το ότι πρόκειται να ακυρώσουμε και τις αναθεωρημένες ε, συμβάσεις της ΔΟΕ τώρα, αλλά όχι μόνο τις της ΔΟΕ. Ε, αν δείτε, αλλά όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της και αν κοιτάξετε τα Ηνωμένα Έθνη θα δείτε ότι σε όλο τον κόσμο εφαρμόζονται οι συμβάσεις αυτές και οι κώδικες διοντολογίας οι παγκοσμίως λοιπόν εφαρμόζονται από όλους τους εμπόρους και γι' αυτό πρέπει το ίδιο να γίνει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή ζητεί από τα κράτη-μέλη να δώσουν το καλό παράδειγμα κυρώνοντας και εφαρμόζοντας τις συμβάσεις αυτές στο ψηφίσμα που ενέκρινε το Μάιο του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είπαμε ότι η ενίσχυση της εφαρμογής και επιβολής του εργατικού δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλων των συμβάσεων της ΔΟΕ πρέπει να είναι προτεραιότητα για τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και τα κράτη-μέλη. Αυτό λοιπόν ε, κάνουμε σήμερα το βράδυ. Ζητούμε από την Προεδρία του Συμβουλίου να είναι όσο φιλόδεξη γίνεται να επιμείνει στα επιχειρήματα τα οποία επιρρονίουν την ανάγκη κύρωσης και εφαρμογή των συμβάσεων αυτών και ζητούμε και από τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τις συμβάσεις αυτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης πρέπει να είναι συνεπής μεταξύ των, της εσωτερικής και της εξωτερικής πολιτικής που εφαρμόζει και να εφαρμόζει και τις βέλτιστες πρακτικές σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα για το πώς μπορούν να εφαρμοστούν οι βέλτιστες πρακτικές και στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό και παγκοσμίω δίνοντας το καλό παράδειγμα σήμερα 26 Νοεμβρίου 7.600 κυρώσεις 600 ε, συμβάσεις περίπου της ΔΟΕ έχουν κυρωθεί ενώ όπως αγωνιζόμαστε για την αλλαγή την κλιματική στην Κοπεχάγη το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εδώ. Ρινό έχει το λόγο για δύο λεπτά παρακαλώ. Ja, tak for ordet. Øh, på vegne af de grønne, så vil jeg gerne understrege, at vi finder bud... Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρου των Πρασίνων θα ήθελα να πω ε, ορισμένα πράγματα για την κύρωση και την εφαρμογή των αναθεωρησμένων συμβάσεων τη ΔΟΕ, που είναι πάρα πολύ απαραίτητη και επίγουσα για δύο λόγους. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να γνωρίζει τι συμβαίνει με την καταπολέμηση της παράνομης εργασίας. Πρέπει να πρωτοστατήσουμε όσον αφορά την δημιουργία καλών συνθήκων εργασίας και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το είπαμε και σήμερα Διαφορετικά θα υπάρχει πολύ μεγάλο χάσμα ανάμεσα σε αυτά που λέμε και σε αυτά που κάνουμε και στις, ε, μεταξύ των εσωτερικών και των εξωτερικών μας σχέσεων. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να αμελήσουν αυτές τις, την κύρωση αυτών των αναθεωρημένων ε, συμφάσεων γιατί θα είχε επιβλαβεί συνέπειες για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για, στις οποίες επίσης συζητούμε να κυρώσουν τις συμβάσεις αυτές. Είναι είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να προηγηθεί, να πρωτοστατήσει σε όλη αυτή τη διαδικασία υπέρ καλών συνθήκων εργασίας και ανταγωνιστικότητας. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Η ΔΟΕ είναι το μέσο που μας δίνει τη δυνατότητα να ε, προχωρήσουμε από κοινού ε, σε διεθνές επίπεδο και πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη η ομάδα των Πρασίνων ε, συμπορεύεται με όλα τα μηνύματα της συγκεκριμένης δήλωσης για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τσίμερ δεν φαίνεται στην αίθουσα και ήθελα να ρωτήσω αν η κυρία Φιγκιουρέδο, που είναι επίσης συντάκτης, ήθελε να πάρει το λόγο τώρα. Συμφωνείτε. Έχετε το λόγο λοιπόν κυρία Φιγκουρέδο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Υποστηρίζουμε την έκκληση που γίνεται προς τα κράτη-μέλη για να λάβουν υπόψη την κοινωνική πτυχή που συνηγορεί υπέρ της επικύρωσης των νέων συμβάσεων. Από το 1919 η ΔΟΕ έχει δείξει αποφασιστικότητα για κάποιους ε, κανόνες στον τομέα της εργασίας, της απασχόλησης, της κοινωνικής ασφάλισης, της, ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με αυτά τα θέματα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είμαστε υπέρ του πρώτου, της πρώτης εκδοχής του ψηφίσματος που εδώ παρουσιάζεται. Δυστυχώς όμως ε, το ΕΛΚ αποφάσισε να μειώσει την ισχύ του ψηφίματος με μια αναφορά στην Λισαβόνα, τη στρατηγική της Λισαβόνας στρατηγική για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Στο όνομα της στρατηγικής της Λισαβόνας είναι η Επιτροπή που παρουσίασε κάποιες από τις χειρότερες προτάσεις για τον εργαζόμενο κόσμο με την ευληγησία, την απορρίθμιση κτλ. Ποιος ξέχασε την οδηγία για το χρόνο εργασίας που απαξιεί τους εργαζομένους, που παρατείνει την ημέρα εργασίας, που θέτει σε αμφισβήτηση τις συλλογικές συμβάσεις και το ρόλο των συνδικάτων. Ακριβώς δηλαδή το αντίθετο από αυτό που πρεσβεύουν οι συμβάσεις της ε, ΔΟΕ. Αυτή η ατυχέστατη αναφορά στη στρατηγική της Λισαβόνας είναι ο λόγος για τον οποίο αποσύραμε την υποστήριξή μας. Στο όνομα όμως της πολιτικής μας ομάδος ζητούμε από τα κράτη-μέλη να επικυρώσουν τις συμβάσεις ε, της Διεθνής, Διεθνούς Οργανώσεως ε, ε, Εργασίας. Ευχαριστώ. Γιουρέδο και τώρα ο κύριος Δεγκούφτο, επίτροπος εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτές, τα τελευταία χρόνια επανειλημμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε την ε, προσήλωσή της στην ε, διεθνώς εγκεκριμένη ε, ημερήσια διάταξη, αν θέλετε, σχετικά με τις συμβάσεις αυτές της ΔΟΕ. Πιστεύουμε ότι ε, οι κυρώσεις αυτές πρέπει να εφαρμόζονται, να εφαρμόζονται φιλόδοξα ε, standards για να μπορέσουν να εφαρμοστούν κανόνες αξιοπρεπούς και δίκαιες ε, εργασίες. Τονίστηκε η ε, σημασία αυτού του προγράμματος εργασίας για αξιοπρεπή εργασία και πιστεύουμε ότι όλες οι κυρώσεις, οι συμβάσεις της ε, ΔΟΕ ε, που αναφέρονται στα διεθνή στάνταρτ πρέπει να κυρωθούν, να εφαρμοθούν, εφαρμοστούν και μέρος της νέας κοινωνικής ε, ατζέντα της ε, Κομισιόν είναι και οι αναθεωρημένες ε, συμβάσεις της ΔΟΕ ζητώντας να κυρωθούν και να εφαρμοστούν όλες ανεξαιρέτως συμβάσεις πιστεύουμε ότι εκπληρούμε έναν ε, σημαντικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποβάλαμε επίσης και προτάσεις για, προς το Συμβούλιο για την ε, ε, όπου ζητούμε να γίνει κύρος και εφαρμογή των αναθεωρημένων συμβάσεων ως το δυνατόν πιο γρήγορα. όπως επίσης και την ε, σύμβαση για την αλία. Ελπίζουμε να ε, γίνει κάτι τέτοιο το, και τα αποτελέσματα θα δημοσιοποιηθούν το 2011. Θα πάρουν το λόγο μιλητέ εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων για την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, ο κύριος Όρη για δύο λεπτά έχει το λόγο. Köszönöm a szót, elnök asszony. Mindenek előtt szeretném üdvözölni a sikerült a frakcióknak megállapodni a nemzetközi munkaügyi. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι που ουσιαστικά όλοι συμφωνούμε ε, μπορέσαμε να συμφωνήσουμε για την κύρωση και την εφαρμογή των αναθεωρημένων συμβάσεων της ΔΟΕ. Η ΔΟΕ είναι μια από τις παλιότερες τις πιο παλιές υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών ιδρύθηκε το 1919 με σκοπό να ορίσει και κανόνες δίκαιης και αξιοπρεπούς δουλειάς για να μην γίνεται εκμετάλλευση των εργαζομένων. Η ε, πολιτική μου ομάδα ε, της ΕΛΚ πιστεύει ότι η τήρηση ορισμένων κανόνων και προτύπων η δημιουργεί τις σωστές συνθήκες και ίσως βοηθήσει να μπορέσουμε να βγούμε και από την οικονομική κρίση στην οποία βρισκόμαστε μέχρι τώρα τα πρότυπα, οι νόρμες ισχύουν και πρέπει να εφαρμόζονται και οι κοινωνικοί εταίροι και οι κυβερνήσει των κρατών μελών πιστεύουμε ότι πρέπει να ε, εγκρίνουν και να εφαρμόσουν όλα τα πρότυπα ε, τα οποία προβλέπονται στις συμβάσεις αυτές. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι εκείνη η οποία ε, κυρώνει τις συμβάσεις της ΔΟΕ. Τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα γι' αυτά βάσει της αρχής επικουρικότητας και ίσως θα πρέπει κάποια στιγμή να συζητηθεί το θέμα αυτό των αρμοδιοτήτων της Ένωσης και των κρατών μελών των ξεχωριστών αρμοδιοτήτων ανάλογα με τα πρότυπα. Μέρος της ε, ε, ομάδας ε, Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για δύο λεπτά ο κύριος Κρίστερσεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Έχουμε μια εσωτερική αγορά, μια ελεύθερη αγορά πολλούμε προϊόντα, υπάρχει ελεύθερος ανταγωνισμός ε, και μπορούμε να αγοράζουμε και φθηνά προϊόντα. Και αυτά όλα πολύ καλά. Αλλά υπάρχουν και άλλα στοιχεία που είναι σημαντικά. Τα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων που πρέπει να εξασφαλίζονται παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν πρέπει να ανταγωνιζόμαστε ως προς αυτό ε, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μειώνοντας τις συνθήκες εργασίας και τους ε, μισθούς. Οπότε μια καλή συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχουμε τις ίδιες αξίες και μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις συμβάσεις ε, της ε, ΔΟΕ για να μπορέσουμε να κινηθούμε προς το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Δυστυχώ τα πράγματα δεν έχουν έτσι ακόμη σήμερα, γιατί προφανώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι είναι υποχρεωτικέ οι συμβάσει ε, μόνο όταν έχουν κυρωθεί από 50% των κρατών μελών. Άρα όλα τα κράτη-μέλη θα έπρεπε να τι ε, κυρώσουν αυτέ τι αναθεωρημένε συμβάσει ε, και που έχουν πλέον καταγραφεί ω τέτοιε. Δεν πρέπει να χάνουμε κι άλλο χρόνο με λόγια. Πρέπει να περάσουμε στην πράξη. Αλλιώ πώ θα ζητήσουμε από άλλε χώρε του κόσμου να κυρώσουν και να εφαρμόσουν τι τις συμβάσεις αυτές. Ε, πώς θα ζητήσουμε από τον ΠΟΕ να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων παντού. Πρέπει να είμαστε εμεί πρώτα υποδειγματικοί. Και τότε θα είμαστε πραγματικά πιστικοί όταν θα ζητούμε από τους άλλους ε, να κυρώσουν τις συμβάσεις. Η αξιοπρεπής εργασία, ναι. Αυτή είναι η απάντηση που πρέπει να δώσουμε στην παγκόσμια κρίση στην οποία διερχόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κρίστορσεν. Και η κυρία Σρέντερ, την ομάδα των Πρασίνων, έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρος. Είναι γεγονός αγαπητοί συνάδελφοι ότι ότι διερχόμαστε μια κρίση και κατά τη διάρκεια κρίσεων ε, πλήττονται συνήθως τα δικαιώματα των εργαζομένων. Πολλές φορές ακούγονται πράγματα ε, σε τέτοιου είδους δυσμενείς συνθήκες ε, που δεν θα έπρεπε να ακούγονται όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση κρίνει τρίτες χώρες, αναφέρεται στην ανάγκη τήρηση ορισμένων βασικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Όμως αυτά παραμένουν λόγια στο εσωτερικό της Ένωσης. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν δικαιώματα τα οποία... Ε, ε, υπάρχουν προβλήματα όπως παραδείγματο χάρη η κατάργηση ουσιαστικά του δικαιώματος της απεργίας σε ορισμένες περιπτώσεις που δεν θα έπρεπε να τα ζούμε το, δι, το ΔΕΚ το δικαστήριο έχει καταγγείλει τέτοιου είδους καταστάσεις κατάλογο των ομιλητών η κυρία έχει το λόγο για δύο λεπτά παρακαλώ Madame Κύριε Πρόεδρε, ε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους του ΕΛΚ αλλά και, της, ε, και των υπολείπων πολιτικών ομάδων γιατί όλοι θελήσαμε γύρω από αυτό το θέμα της αξιοπρεπούς εργασίας να συμφωνήσουμε για να υποβάλουμε ένα κοινό ψήφισμα και οι διαπραγματεύσεις των τελευταίων ημερών ήταν πάρα πολύ θετικές. Από το 1919 η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας μπόρεσε να εξασφαλίσει και να αναπτύξει ένα σύστημα κανόνων, διεθνών κανόνων για την εργασία που καλύπτουν ε, ένα μεγάλο πρίσμα ε, ζητημάτων όπως η κοινωνική πολιτική, η εργασία, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν μπορούμε να το ξεχνούμε, δεν μπορούμε να το, να το παραγνωρίζουμε, ειδικότερα σε μια περίοδο κρίσεως. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όλες αυτές οι συμβάσεις ε, που θεωρήθηκαν πλέον αναθεωρημένες κατόπιν μιας τριμερής διαδικασίας και που ε, συνδέουν ε, τους εργοδότες, τους και τις κυβερνήσεις. Γι' αυτό ακριβώς εμείς κάναμε αυτή την έκκληση, αυτή τη σύσταση στα κράτη-μέλη, ζητώντας τους να κυρώσουν αυτές τις συμβάσεις, ζητώντας τους να συνεισφέρουν στην πραγματική εφαρμογή τους για την εξέλιξη για την ανάπτυξη της κοινωνικής Ευρώπης. Θέλουμε λοιπόν ε, σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα επαγρυπνήσουμε όσον αφορά την, ε, το σεβασμό των προθεσμιών αυτών ε, να εφαρμοστούν οι συμβάσεις αυτές με το σεβασμό της επικουρικότητας. Η ομάδα του ΕΛΚ θα είναι ιδιαίτερος προσεκτική για την εφαρμογή των συμβάσεων στα κράτη-μέλη, κατα της παράνομης εργασίας, την, το κοινωνικό μοντέλο και την πρακτική πραγματική ε, κοινωνική Ευρώπη που ε, θα δείξει το σωστό δρόμο σε όλο τον κόσμο και θέλουμε πραγματικά να υπάρξει εξέλιξη προς αυτήν την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα το λόγο θα πάρει η κυρία Ράπτη για δύο λεπτά επίσης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μία από τις σημαντικές ιδιαιτερότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η σημασία που αποδίδει στην κοινωνική πολιτική και στα θεμελιώδη δικαιώματα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η εφαρμογή των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει ένα κράτος μέλος της Ένωσης. Όπως ξέρουμε ότι τα δικαιώματα αυτά όταν καταπατούνται δημιουργούν στην Ένωση την υποχρέωση να επιβάλλει κυρώσεις. Η σύμφυτη με τη δημιουργία και λειτουργία της Ένωσης θεμελίωση των δικαιωμάτων αυτών επεκτείνεται και στον εργασιακό χώρο. Η σημασία που η Ένωση αποδίδει στην προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων δεν είναι εμφανή μόνο όταν παράγεται εσωτερική νομοθεσία, αλλά και στην εξωτερική τη πολιτική. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όταν πρόκειται να κάνει συμβάσει με τρίτε χώρε, μία από τι προποθέσει που θέτει είναι να γίνονται σεβαστά, τα βασικά εργασιακά δικαιώματα. Για αυτού του λόγου, η Ένωση δεν θα μπορούσε παρά να είναι από του προτεργάστε για τη στήριξη και την αναγκαία συστηματική αναθεώρηση των συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας της ΔΟΕ. Πρόσφατα, μετά από διαπραγματεύσεις με εργαζόμενους, εργοδότες και με τις κυβερνήσεις, η ΔΟΕ προχώρησε σε μια ακόμη αναθεώρηση των συμβάσεών της. Και ενώ οι κυβερνήσεις των κρατών μελών, αλλά και η Ένωση, είναι ανάμεσα σε όσους συμμετείχαν στην εν λόγω αναθεώρηση, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα παράδοξο το παράδοξο αυτό είναι ότι πολλά κράτη-μέλη της Ένωσης, ενώ έχουν υιοθετήσει ενωσιακές οδηγίες που επιβάλλουν εργασιακά δικαιώματα πιο προωθημένα από αυτά των συμβάσεων της ΔΟΕ, υποτιμούν τη σημασία του τυπικού ζητήματος να κυρώσουν σε εθνικό επίπεδο τις συμβάσεις αυτές. Επειδή η εικόνα που δίνουμε με τον τρόπο αυτό προς τρίτες χώρες και μάλιστα προς αναπτυσσόμενες χώρες είναι στρεβλή, θα είναι εύλογο να αλλάξουμε νοοτροπία και να προχωρήσουν τα κράτη-μέλη όσα δεν το έχουν κάνει στις απαραίτητες κυρώσεις. Και εν πάση περιπτώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κύριε Επίτροπε, ας μην διστάζει να ζητά πιο δυναμικά από τα κράτη-μέλη να εκπληρώνει τέτοιες υποχρεώσεις, ώστε να αυξηθεί η αξιοπιστία της Ένωσης με την πρόθεση της αξιοπρεπούς εργασίας, ιδιαίτερα μάλιστα στην σημερινή συγκυρία της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Εμβόλυμα θα πάρει το λόγο ο κύριος Λεϊαρίκ για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, προφανώς και πρέπει να επιμείνουμε για να εφαρμοστούν οι συμβάσεις ε, της ΔΟΕ. Φοβούμε όμως ότι το σύστημα αυτό το οποίο έχουμε επιλέξει του ελεύθερου ανταγωνισμού θα καταστήσει, για να μην πω θα καταντήσει, την εργασία ένα εμπορικό αγαθό. Θέλουμε ε, αυτές οι απειλές και οι πιέσεις να μην ε, υφίστανται. Υπάρχει ένα παράδειγμα στη Γαλλία. Μία επιχείρηση ε, έκλεισε για να μετακατεσταθεί στη Βουλγαρία και ζητούμε από αυτή την, από την επιχείρηση να πάει να καταρτήσει να μάθει δηλαδή τη δουλειά στους βούλγαρους εργαζομένους. Αυτή είναι η πολιτική που οδηγεί στην μεταγκατάσταση, στις πιέσεις που υφίστανται οι εργαζόμενοι και στην υποχώρηση των κοινωνικών προτύπων. Θα πρέπει να εξευρεθεί ένα σύστημα εναρμόνισης προς τα πάνω των κοινωνικών συστημάτων, ούτω ώστε να μην υπάρχει πια αυτός ο ανταγωνισμός, ο αδυσόπιτος ανταγωνισμός ε, μεταξύ των επιχειρήσεων και άρα μεταξύ των ίδιων των εργαζομένων. Ομοίως δεν θα πρέπει να συνεχίσουμε να προχωρούμε προς αυτό που ονομάζουμε και εδώ και στην Κομισιόν Flexicurity, ευελισφάλεια αλλά προς ένα σύστημα επαγγελματικής κοινωνικής ασφάλισης που να συνδυάζεται με περίοδους κατάρτισης και εκπαίδευσης που είναι πάντα απαραίτητες. Έτσι μόνο θα διέλθουμε τις κρίσεις, έτσι θα εκπαιδεύσουμε τους εργαζομένους, έτσι θα τους κατορτήσουμε, έτσι θα τους βοηθήσουμε να οδηγηθούν προς τις δουλειές, τα επαγγέλματα που πρέπει να εφεύρουμε για το μέλλον ήθελα να σας ε, εξηγήσω ότι ο κύριος Ιαρίκ δεν πήρε το λόγο, τον πήρε εμβόλυμα, αλλά όχι τυχαία. Αντικατέστησε την κυρία Φιγκιουρέδο, η οποία αντικατέστησε την κυρία Τσίμερ. Το λέω για να μην έχουμε τήσεις εμβόλυμων παρεμβάσεων. Τώρα το λόγο θα πάρει για 1,5 λεπτό ο κύριος Λούβινγκσον. Mr. Ja, fru talman. E έχει εγκριθεί η συνθήκη της Λισαβόνας, το γνωρίζουμε. Τα... Η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων έχει επίσης εγκριθεί. Και σήμερα έχουμε μία νέα δυνατότητα που ανοίγεται για την ε, κοινωνική Ευρώπη. Ένα πρώτο καλό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή θα είναι η κύρωση το συντομότερο δυνατόν όλων των αναθεωρημένων συμβάσεων ε, της ε, ΔΟΕ. Υπάρχει επίσης και μια εξωτερική πτυχή. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να είναι ένα σοβαρό εταίρο ε, στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας για την βελτίωση των συνθήκων εργασίας και διαβίωσης, είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη να εγκρίνουν τις σχετικές συμβάσεις. Και αν θέλουμε να ασκήσουμε επιρροή σε τρίτες χώρες, πρέπει να ξεκινήσουμε δίνοντας το καλό παράδειγμα. Οπότε κάνω έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προς τη Σουηδική Προεδρία. Θα ήθελα να είμαστε πιο προοδευτικοί, να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο ώστε όλες αυτές οι αναθεωρημένες συμβάσεις να γίνουν αποδεκτές από όλα τα κράτη-μέλη. Βεβαίως και η δική μου χώρα, ε, η Σουηδία, δεν έχει ακόμη ε, κυρώσει σημαντικές ε, συμβάσεις, όπως για παράδειγμα αυτή του 96 για τις δημόσιες συμβάσεις. Πραγματικά λυπούμε πάρα πολύ γι' αυτό και θα ήθελα η, Διεθνή, η Σουηδική Προεδρία να κάνει όσο ό,τι μπορεί για να γίνει αυτό στο δυνατόν περισσότερα. Θα ήθελα λοιπόν όλα αυτά να καταστούν υποχρεωτικά και τότε μόνο το ΔΕΚ θα έχει λιγότερη δουλειά. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε μια κατάσταση κατά την οποία από τη μία έχουμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία η οποία δεν λαμβάνει υπόψη τις συμβάσεις της ΔΟΕ. Ε, για, είμαστε στη διαδικασία Catch the Eye. Για ένα λεπτό μπορούν να πάρουν το λόγο οι συνάδελφοι που έχουν ζητήσει. Ε, πρώτη έχει ζητήσει το λόγο η κυρία Μακκίνες. Έχετε το λόγο, κυρία συνάδελφε, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Εδώ, όπως είπαν οι συνάδελφοι, από το 1919 δραστηριοποιείται στον τομέα 90 χρόνια και ακόμα εργάζεται ε, για το θεματολόγιο τη αξιοπρεπού εργασία. Είναι πολύ σημαντικό τα κρατημέλη, όπω είπαν και άλλοι, να επικυρώσουν όλε τι κυρώσει, ιδιαίτερα στη στιγμή τη κοινωνική και κυρίω οικονομική κρίση που διερχόμεθα. Γι' αυτό ακριβώ θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το ρόλο της ΔΟΕ στον ε, αναπτυσσόμενο κόσμο, την συνεργασία του με τις ε, ΜΚΟ, ιδιαίτερα για την προστασία των πιο ευάλωτων, των αναπήρων α πούμε, που ποτέ δεν θα είχαν καμία ευκαιρία αν δεν υπήρχαν αυτά τα προγράμματα. Είναι και άλλοι πολύ σημαντικοί τομείς, ε, η παιδική εργασία, η σκλαβιά, και αν ε, το καταφέρουμε αυτό, ε, αν θέλουμε να το καταφέρουμε, το ελάχιστο που πρέπει να κάνουν τα κρατημέλη είναι να επικυρώσουν πλήρως όλες τις συμβάσεις για να δώσουν το καλό παράδειγμα. Ευχαριστώ. Κύριε Μακίνες, ο κύριος Σιεκέρσκι έχει ζητήσει επίσης το λόγο. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Międzynarodowa Organizacja Pracy w ciągu wielu lat swojej działalności przyjęła i przedstawiła do Σε όλα τα χρόνια της λειτουργίας της ΙΔΟΕ έχει προτείνει πολλές διεθνείς συμβάσεις ε, και οδηγίες που έχουν να κάνουν με την εργασία, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθε, τα συνδικάτα και την κοινωνική ασφάλεια, όπως επίσης και τις συνθήκες εργασίας. Τα κράτη-μέλη πρέπει να κυρώσουν και να σεβαστούν τις εν λόγω συμβάσεις. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επίσης να συμβάλλει σε ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως είναι η προστασία των ε, δικαιωμάτων των εργαζομένων σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Κάθε πολίτης πρέπει να εξασφαλίσουμε ε, κάθε πολίτης οποιασδήποτε φυλής, οποιασδήποτε προτίμησης πρέπει να προστατεύεται και να έχει τη δυνατότητα ε, οικονομικής ασφάλειας και ίσων ευκαιριών. Η ένδια, ανεξαρτήτως του που υπάρχει, είναι μια πολύ μεγάλη απειλή. Έχει άλλος συνάδελφος ή συνάδελφος Και παρέμβει. Δεν βλέπω να είναι αυτή η περίπτωση, οπότε ο κύριος Επίτροπος έχει και πάλι το λόγο. Ε, Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχει σύγκληση απόψεων για την ανάγκη να κυρωθούν και να εφαρμοστούν οι συμβάσεις της ΔΟΕ όπου συμφωνεί λοιπόν και το Κοινοβουλίο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά όπως ε, είπε και ο κ. Σωρή υπάρχουν ε, κάποιες αρμοδιότητες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να επιβάλλει ορισμένα πράγματα σε ορισμένες περιπτώσεις αλλά όχι σε άλλες. Η, το, το ΔΕΚ αναγνωρίζει ως ανθεμελιώδες δικαίωμα την ε, μαζική διαδήλωση αν θέλετε ή τη μαζική συνδικαλιστική δράση. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δεχτούμε. Και όπως είπαμε και πριν βεβαίως η συμβάση της ΔΟ είναι μέρος της βασικής κοινωνικής πολιτικής μας. Κληρώνοντας τη συζήτηση αυτή θέλω να σας αναγγείλω ότι έχω λάβει τρεις προτάσεις ψηφίσματος. Η μία πρόταση είναι από κοινού από την ε, ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και την ομάδα των Φιλελευθέρων με την ομάδα της Αριστεράς. Η άλλη πρόταση είναι